Να συνεχίσουμε λοιπόν τις εργασίες μας από το σημείο 27 στην ημερήσια διάταξη. Δικαιώματα των επιβατών, λεωφορείων και πούλμαν. Ε, εισηγητής ο κύριος Γκαμπριέλ Αλμπερτίνη. Θα εξετάσουμε το σχέδιο ε, έκθεσης. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Με αυτή την πρόταση για τα δικαιώματα των επιβατών ε, λεωφορείων και πούλμαν, η Ευρωπαϊκή Ένωση συμπληρώνει το νομοθετικό πλαίσιο για όλα τα μέσα μεταφοράς. Να σας υπενθυμίσω την πρόσφατη έγκριση της νομοθεσίας για τις εναέριες μεταφορές, ε, το οποίο θα διορθώσουμε στο μέλλον, και φυσικά τις σιδηροδρομικές μεταφορές, για να μην ξεχνάμε και αυτό το οποίο θα συζητήσουμε σήμερα το απόγευμα, την έκθεση του συναδέλφου Ντεσενέ για τις ε, θαλάσσιες μεταφορές και τις εσωτερικές ε, οδούς ναυσιπλοείας. Ε, εξετάζοντας αρχικά το θέμα αυτό, θεώρησα ότι υπήρχε ανάγκη να βρεθεί μια ισορροπία μεταξύ δύο εξίσου σημαντικών ε, ε αναγκών αλλά κατά πάσα πιθανότητα αντιφατικών. Ε, αφενός έπρεπε να έχουμε ένα νομοθετικό πλαίσιο, το λεγόμενο level playing field, το οποίο θα επιτρέπει σε όλα τα διάφορα μέσα μεταφοράς να είναι ανταγωνιστικά μεταξύ των ε, με τις ίδιες ευκαιρίες και με ίσες ευκαιρίες και με, ταυτόχρονα να έχουν οι επιβάτες τα ίδια δικαιώματα και το ίδιο υψηλό επίπεδο προστασίας ανεξάρτητα από το μέσο μεταφοράς το οποίο θα έχουν επιλέξει. Το νομοθετικό πλαίσιο βέβαια, πέρα από αυτή την ε, γενικότερη ε, ιδέα των πραγμάτων θα πρέπει να αντικατοπτρίζει και τις ιδιαιτερότητες ε, και τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά ε, του κάθε μέσου μεταφοράς. Να σας κάνω ένα παράδειγμα για να γίνω κατανοητός. Είναι τελείως διαφορετική η διαχείριση των καθυστερήσεων σε περίπτωση ε, μεταφοράς ε, με αυτοκίνητο όχημο που χρησιμοποιεί τους δρόμους ε, για τις δημόσιες μεταφορές με τα ΙΟΤΑΧΗ που σημαίνει ότι ε, μπορεί να υπάρχουν ατυχήματα, μπορεί να υπάρχουν αρκετές ε, περιπτώσεις που μπορεί να οδηγήσουν σε καθυστέρηση ε, σε σχέση με τα όσα έχουμε στο σιδηρόδρομο που υπάρχει μια συγκεκριμένη οδός η οποία είναι ad hoc ανατεθειμένη στο σιδηρόδρομο, στο τρένο. Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους συνεργάστηκαν μαζί μου σε αυτή την προκαταρκτική φάση, διότι επέδειξαν μεγάλη δέσμευση προς το θέμα και μεγάλη ικανότητα εργασίας, διότι η προθεσμία για το σχέδιο έξεσης ήταν πάρα πολύ μικρή και δεν υπήρξε δυνατότητα Συγγνώμη, υπήρξε δυνατότητα να συναντήσουμε και τους εκπροσώπους των μέσω μαζικής μεταφοράς, ε, όπως επίσης και τους ε, εκπροσώπους των επιβατών και ατόμων με κάποια αναπηρία ή με κάποια δυσκολία στη μετακίνηση. Μίλησα επίσης και με το Προεδρείο του ε, Επιτρόπου Αρμόδιου για τις Μεταφορές και την Ενέργεια. Και στις επόμενες ημέρες θα δούμε τα εκκρεμή ακόμα θέματα με τους σκιώδεις εισηγητές από τις διάφορες πολιτικές ομάδες από τις επόμενες ώρες θα συναντηθώ με τους πρώτους εξ αυτών. Πριν να αφήσω λοιπόν το λόγο στους συναδέλφους για να ξεκινήσουμε τη συζήτηση, θα ήθελα να σταθώ εν συντομία σε κάποιες τροποποίησεις που παρουσίασα στο σχέδιο έκθεσης και που θεωρώ ότι είναι ιδιαίτερα ουσιαστικές. Και θα πρέπει να τις επισημάνω εδώ. Αναφέρομαι στις τροπολογίες 3, 7, 19 και 20, οι οποίες αφορούν μία σειρά από άρθρα τα οποία φρονώ ότι θα πρέπει να εμβαθύνουμε με ιδιαίτερη προσοχή. Επιφυλάσσομαι λοιπόν για να παρουσιάσω και ίσως ε, κάποιες περαιτέρω διορθώσεις επί των άθρων αυτών και αφότου θα έχω ακούσει την άποψη, την έγκυρη φυσικά και τα σχόλια τα οποία θα προκύψουν από τους συναδέλφους, ε, καταρχάς ε, από τους κοιόδης εισηγητές που όπως σας είπα θα συναντήσω ακόμα και μέσα στις επόμενες λίγες ώρες. Σε αυτά τα σημεία, για να εμβαθύνουμε, θα επανέλθω σε λιγάκι. Κάποιες διευκρινήσεις για τις τροπολογίες 4, 5 και 6. Εδώ ε, προτείνω να διορθώσουμε κάποιους από τους ορισμούς που αναφέρουμε στο άρθρο 3, πιο συγκεκριμένα τη σύμβαση μεταφοράς, το εκδοτήριο εισιτηρίων και τον ταξιδιωτικό πράκτορα. Επίσης, στο άρθρο 11 για τις ε, παρεκκλήσεις και τις ειδικέ ε, προϋποθέσεις ήθελα να έχω κάποιες διευκρινιστικές τροπολογίες, πιο συγκεκριμένα τις 8, 9, 10 και 11. Να σταθώ στην ε, τροπολογία 8, στην οποία λαμβάνω υπόψη το γεγονός ότι μέχρι τούδε δεν υπάρχει ενισχύ νομοθεσία τόσο τοπική όσο εθνική και ευρωπαϊκή που να επιτρέπει σε μία επιχείρηση η οποία παρέχει υπηρεσίες ε, μεταφοράς μέσω λεωφορείων ή πούλμαν να περιορίσει την ε, ε, μεταφορά ατόμων με αναπηρία για λόγους ασφαλείας. Οι τροπολογίες 12, 13, 21 και 22 είναι απλά διευκρινιστικές οι οποίες όμως πιστεύω ότι είναι απαραίτητες και μου τις ζήτησαν οι οργανώσεις ατόμων με αναπηρία ή με περιορισμένη κινητικότητα και αφορούν την ε, έννοια του ε, accessible format. Επίσης, ε, προσπάθησα να βρω και μία συμβιβαστική λύση μεταξύ του αιτήματο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που προέβλεπε ένα χρόνο για τη θέση σε ισχύ του κανονισμού και την ε, θέση που μας ε, εξέφρασαν ε, οι φορείς του κλάδου, οι οποίοι θεωρούν ότι για να προσαρμοστούν στις νέες απαιτήσει του κανονισμού χρειάζονται τρία χρόνια. Στον, στην τροπολογία λοιπόν τη σχετική είμαι κάπου ανάμεσα στις δύο, μια μέση λύση. να επανέλθω τώρα εν συντομία σε κάποιες βασικές τροπολογίες, πιο ουσιαστικές, ε, θέματα στα οποία θεωρώ ότι θα πρέπει να σταθούμε λίγο περισσότερο για να μπορέσουμε να συζητήσουμε και σήμερα και να φτάσουμε σε πιο κατάλληλους ορισμούς. Ε, αναφέρομαι καταρχάς στο άρθρο 2.2 που αφορά στο πεδίο εφαρμογή. Εδώ θα πρέπει να διασφαλίσουμε Αφενός ότι θα έχουμε ένα επίπεδο προστασίας για τους επιβάτες λεωφορείων και πούλμαν παρόμοιο με αυτό το οποίο αναφέρεται στον κανονισμό, δηλαδή ε, το obligation de resultat. Επίσης θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και την συγκεκριμένη ιδιαιτερότητα των αστικών ε, και τοπικών συγκοινωνιών. Επομένως θα πρέπει να δούμε και τι γίνεται με την εφαρμογή αυτού του κανονισμού με συγκεκριμένη αναφορά σε αυτό το τομέα. Και επίσης υπάρχει το άρθρο 6 που αφορά την ευθύνη σε περίπτωση ε, ε, ατυχήματος ή ε, τραυματισμού των επιβατών. Για το θέμα αυτό είμαστε σε επαφή με τους ε, εκπροσώπους των ασφαλιστικών εταιριών καθώς επίσης και τους υπαλλήλους της Γενικής Διεύθυνσης Τρέν και Εσωτερικής Αγοράς και φυσικά με το, προεδρείο, με το γραφείο του Επιτρόπου Ταγιάννη για να καταλήξουμε σε μια κοινά αποδεκτή λύση. Τέλος, το άρθρο 20 που αφορά στην ευθύνη σε περίπτωση ακύρωσης ή παρατεταμένης καθυστέρησης. Εδώ νομίζω ότι το κείμενο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής χρήζει κάποιον περαιτέρω διευκρινήσεων προκειμένου να είναι πιο σαφές και πολύ πιο εύκολο στην ερμηνεία του. Ε, θεωρώ ότι εδώ θα πρέπει να καταθέσω και κάποιες επιπλέον τροπολογίες ε, όσον αφορά στον ορισμό της καθυστέρησης ε, και την υπόθεση που χρησιμοποιεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που προβλέπει για την περίπτωση αποζημίωσης καθυστερήσεις άνω των δύο ερών για ταξίδια άνω των τριών ωρών, ε, διότι θεωρώ ότι αυτό είναι πολύ περιοριστικό. Τώρα, για τις υποχρεώσεις των ε, ε, μεταφορικών εταιριών, ε, για παράδειγμα κάποια γεύματα ή κάποια παραμονή σε ξενοδοχείο, ε, τα οποία δεν προβλέπονται προς το παρόν. Εγώ δεν έχω κάτι άλλο να προσθέσω, έχω τα αυτιά μου τεντωμένα λοιπόν, τίνω ευήκο για να ακούσω τι έχετε να μου πείτε και ελπίζω να μου ε, δώσετε τις παρατηρήσεις σας, διότι όπως σας είπα σε κάποια από αυτά τα θέματα χρειάζομαι τη συνεργασία σας για να μπορέσω να πλαισιώσω λίγο καλύτερα την έννοια του θέματος και τα όσα προκύπτουν από αυτόν τον κανονισμό σας. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε τον κύριο ε, Αλμπερτίνη, ο κύριο Εύανς. Thank uh, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον κύριο Αλμπερτίνη για την παρουσίαση που μας έκανε. Συγγνώμη για την καθυστέρηση επίσης. Έχασα λίγο την αρχή της παρεμβασής του. Πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντική η έκθεση αυτή, το νομοθέτημα αυτό, εγώ ήμουν εισηγητή για την πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία και μειωμένη κινητικότητα στα αεροπλάνα, σε μια έκθεση που εξετάσαμε πριν από μερικά χρόνια και είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένο προσπαθούμε αυτή τη φορά να επεκτείνουμε το πεδίο εφαρμογή αυτού του καονισμού στους επιβάτες λεωφορείων και πούλμαν και θεωρώ ότι θα δώσουμε κατά αυτόν τον τρόπο ένα πολύ θετικό μήνυμα προς Ευρωπαίους πολίτες, ιδίως πριν από τις ευρωπαϊκές εκλογές. Θεωρώ το μαθέτημα αυτό θα ωφελήσει εκατομμύρια, θα έλεγα, Ευρωπαίων πολιτών που χρησιμοποιούν λεωφορεία και πούλμαν. Ορισμένες από τις παρατηρήσεις που θα κάνουν ενδεχομένω να ενδιαφέρουν περισσότερο τους κατοίκους του Ηνωμένου Βασιλείου. Ναι, έτσι ήθιστε συνήθως και φαντάζομαι ότι και εσείς ενδεχομένως να επικεντρώνεστε περισσότερο σε θέματα τα οποία αφορούν τη Γερμανία, είναι γερμανικού ενδιαφέροντος, έτσι δεν είναι. Ας συνεχίσουμε όμως. Μα σκέφτομαι ευρωπαϊκά κύριε Πρόεδρε, αλλά εκτός μικροφώνου η παρέμβαση του Πρόεδρου. Λοιπόν, η πρόταση αυτή αφορά τις εσωτερικές αλλά και διεθνείς μεταφορές με λεωφορεία και πούλμαν και θα πρέπει να καταστήσουμε απόλυτα σαφές σε ποιο επίπεδο θέλουμε να εφαρμοστεί το νομοθέτημα αυτό. Στα αγγλικά χρησιμοποιείται ο όρος bus, πράγμα το οποίο σημαίνει κάτι διαφορετικό από τον όρο coach. Συνήθως η μεταφορά που γίνεται με μπας, δηλαδή λεωφορείο, είναι μια μεταφορά που καλύπτει 30-50 χιλιόμετρα το πολύ. Είναι ουσιαστικά αστική και υπεραστική μεταφορά, ενώ coach, pullman, είναι ένας όρος που αναφέρεται σε μεταφορές πολύ πιο μακρινές, πολύ πιο μεγάλες. Ξέρω ότι οι Αμερικάνοι χρησιμοποιούν τους όρους αυτούς διαφορετικά. Πολλές φορές όταν οι Αμερικάνοι λένε bus journey αναφέρονται ένα πολύ μεγάλο ταξίδι. Θα προσπαθήσω να είμαι προσεκτικός λοιπόν με την ορολογία που χρησιμοποιώ κύριε Πρόεδρε. Στα αγγλικά που μιλάει κανείς στην Αγγλία, όταν λέγεται bus journey εννοούμε ένα ταξίδι πολύ πιο σύντομο, πολύ πιο μικρό. Επομένως θα πρέπει να είμαστε σίγουροι για την ορολογία που χρησιμοποιούμε και πώς θέλουμε να εφαρμοστεί. Τώρα, θα πρέπει να γνωρίσουμε ότι ε, τα λεωφορεία ιδίω συνήθως έχουν μόνο ένα άτομο, τον οδηγό, ως προσωπικό. Θα πρέπει λοιπόν να συνειδητοποιήσουμε ότι καθότι πρόκειται για ένα μόνο άτομο θα πρέπει αυτό να είναι σε θέση να εκτελέσει τα καθήκοντά του, ότι έχει λάβει τη σωστή ε, κατάρτιση, ότι γνωρίζει πώς να αντιμετωπίσει άτομα με μειωμένη κινητικότητα ή άτομα με αναπερίες και ότι θα είναι σε θέση να παράσχει αυτή τη συνδρομή. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι οι υποχρεώσει εδώ πέρα και τα καθήκοντα θα πρέπει να διαφέρουν από οι συνθήκε τουλάχιστον διαφέρουν σε σχέση με τον αεροπορικό τομέα, καθότι εκεί πέρα έχουμε ένα προσωπικό που τελείται από πολλά άτομα. Σε ένα αεροπλάνο έχουμε ε, πολλούς υπαλλήλου ενώ σε ένα πούλμαν ή ένα λεωφορείο, κυρίως ένα λεωφορείο, έχουμε μόνο ένα εργαζόμενο και αυτός είναι ο οδηγός. Τώρα, όσον αφορά ταξίδια με τα πούλμαν, εδώ ενδεχομένω, ακριβώ επειδή το ταξίδι είναι πολύ πιο μεγάλο, να έχουμε δύο οδηγού ή να έχουμε έναν οδηγό και έναν συνοδηγό. Και το άτομο αυτό, το δεύτερο δηλαδή άτομο, εφόσον έχει λάβει σωστή κατάρτιση, θα μπορεί και αυτό με τη σειρά του να παράσχει τι απαραίτητε υπηρεσίε. Επίση, θα πρέπει να διευκρινίσουμε ότι μιλάμε εδώ πέρα για ανταγωνισμό και ορισμένα από ταξίδια τα οποία γίνονται με πούλμαν, τα μεγάλα δηλαδή ταξίδια, έρχονται σε άμεσο ανταγωνισμό με τα τρένα. Και Ορισμένε φορέ συνταγωνισμό επίση και με τα αεροπλάνα, καθότι ενδεχομένω η μεταφορά ανάμεσα σε δύο ευρωπαϊκέ πόλει με πούλμαν είναι πιο γρήγορα από τη μεταφορά με αεροπλάνο. Να αναφερθώ και σε κάτι ακόμα, το οποίο έχει πάλι ένα βρετανικό-αγγλικό χαρακτήρα, αν θέλετε. Είναι ότι Τη δεκαετία του 1980 στην Βρετανία είχαμε πολλά μεγάλα μονοπόλια, μεγάλες βρετανικές εταιρείες ε, λεωφορείων Πούλμαν, οι οποίες διασπάστηκαν σε πολλές μικρότερες εταιρείες στη συνέχεια με τη μεταρρύθμιση του τομέα. Θα πρέπει λοιπόν να γνωρίζουμε ότι έχουμε καταλήξει πολλέ φορέ με εταιρείε οι οποίε διαχειρίζονται μόνο 4 5 λεωφορεία. Θα πρέπει λοιπόν το επίπεδο ευθύνη με το οποίο επιθυμούμε να βαρύνουμε τι εταιρείε αυτέ να είναι ρεαλιστικό. Όταν λέμε λοιπόν ότι κάθε εταιρεία θα πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες της, θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι είναι σε θέση οι εταιρείε αυτές να λάβουν τις ευθύνες οι οποίες εμείς ε, θέτουμε. Καταλαβαίνετε ότι σε πολλές περιπτώσεις μιλάμε για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις ε, για τις οποίες θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι θα είναι όντως σε θέση να αναλάβουν την ευθύνη την οποία περιγράφουμε εδώ πέρα σε αυτή την ε, έκθεση. Πάντως αυτό το οποίο λέει ο κύριος Αλμπερτίνη στην έκθεσή του είναι πάρα πολύ σημαντικό πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές για όλους τους επιβάτες ανεξάρτητα από τη χώρα στην οποία κατοικούν αν θέλουμε πραγματικά να έχουμε μία ενιαία κοινή αγορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η αγορά αυτή δεν θα πρέπει να έχει να κάνει μόνο με προϊόντα και κεφάλαια, αλλά θα πρέπει πραγματικά να είναι σε θέση να ωφελήσει τους Ευρωπαίους πολίτες, τους απλούς πολίτες, οι οποίοι επιθυμούν να κυκλοφορήσουν ελεύθερα και άνετα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είτε πρόκειται με αεροπλάνο, είτε πρόκειται με τρένο, είτε πρόκειται με λεωφορεία ή πούλμαν. Και θεωρώ ότι το νομοθέτημα αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και ελπίζω ότι θα καταφέρουμε πριν από τις εκλογές να ολοκληρώσουμε την ε, εξέταση του εγγράφου αυτού και να καταφέρουμε κατά αυτόν τον τρόπο να φτάσουμε και στις ευρωπαϊκές εκλογές έχοντας κλείσει αυτό το ντοσιέ. Ευχαριστώ. Ε, Ευχαριστώ κύριο Φεράρι. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω τον συνάδελφο Αλμπερτίνη για την έκθεσή του. Μπορούμε κάλλιστα να πούμε ότι πρόκειται για μια πολύ ισορροπημένη έκθεση που αντιμετωπίζει με πολύ καλό τρόπο τα δικαιώματα των εφηβατών. Δέχομαι την πρόταση να κάνουμε κάποιες εξαιρίσεις για τις τοπικές μεταφοράς σε σχέση με τα ε, διεθνή ταξίδια, δεδομένες και τις ιδιωτερότητες, χωρίς βέβαια να υπονομεύσουμε και την ποιότητα της ίδιας υπηρεσίας. Η μόνη μου ανησυχία είναι η τροπολογία 10 που αναφέρεται η περίπτωση του αναπήρου ατόμου στο οποίο έχει αρνηθεί η επιβίβαση λόγω της αναπηρίας του. Συμφωνώ με την τροπολογία του εισηγητή, αλλά δεν θα ήθελα να καταχραστούμε το μέσο της αποζημίωσης του εισιτηρίου ως ε, δικαιολογία ε, διότι δεν διαθέτουμε σε άτομα με συγκεκριμένη αναπηρία ειδικά μέσα μεταφοράς. Επίσης ε, πιστεύω ότι θα πρέπει να έχουμε ένα συγκεκριμένο διάστημα για να προσαρμοστεί κάποιο στον κανονισμό. Κατανοώ ότι αυτά που ζητάει ο κλάδος είναι σωστά, αλλά καταλαβαίνετε ότι οι χρόνοι που δίνονται είναι κατάλληλοι για να προσαρμοστούν στην πρόταση αυτή. Θα ήθελα να διατηρήσουμε την άποψη του κειμένου και ίσως ε, να ε, λάβουμε υπόψη μας σοβαρά και κάποιες από τις προτάσεις του κανονισμού. Ευχαριστώ πολύ κυρία ευχαριστώ πολύ. Θεωρώ ότι είναι πραγματικά πάρα πολύ σημαντικός αυτός ο φάκελος και το λάβαμε καθυστερημένα. Νομίζω ότι σε τελική ανάλυση θα έπρεπε να έχουμε πετύχει στην Ευρώπη να μην υπάρχουν διακρίσεις στις μεταφορές για τα άτομα με αναπηρία και εδώ πέρα υπάρχουν τεράστιες διαφορές μεταξύ των κρατών μελών. Αυτό να το τονίσουμε οι Βρετανοί και οι Βορειοευρωπαίοι μας ξεπερνούν κατά πολύ. Εγώ μιλάω ως κεντρική Ευρώπη. Ναι, ναι, ναι, συνάδελφε Γιαζεμπόσκη. Νομίζω ότι θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε το εξής. Στόχος μας πρέπει να είναι να μην υπάρχει καθόλου διάκριση, να μην υπάρχουν καθόλου διακρίσεις για τα άτομα με περιορισμένες κινητικές δυνατότητες. Αλλά φυσικά θα πρέπει να διαπιστώσουμε ότι θα έρθουμε αντιμέτωποι με αναδιαμορφώσεις, για παράδειγμα πόσο θα πρέπει να αλλάξουν οι στάσεις στα λεωφορεία, αλλά και πώς θα πρέπει να αλλάξουν τα ίδια τα λεωφορεία και οι στάσεις των και τα λεωφορεία θα πρέπει να πετύχουμε την κατάργηση των διακρίσεων. Γιατί όλο και πιο πολλά θα είναι τα άτομα στο μέλλον που δεν θα έχουν ιδιωτικό όχημα, αλλά που θα έχουν δικαίωμα να μετακινηθούν. Και όποιος έχει πάρει ποτέ στη ζωή του παιδικό καρατσάκι για να μετακινηθεί με λεωφορείο ή με τρένο, ξέρει τι περνάει ο ανάπηρος με το αναπηρικό καροτσάκι. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν αυτό. Αν θέλουμε να είμαστε δίκαιοι. Αλλά για το σκοπό αυτό χρειαζόμαστε και καταρχάς πολύ συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα. Τι θα πρέπει να γίνει και μέχρι πότε. Θεωρώ ότι χρειάζονται επίσης πιο σκληρά μέτρα σε ό,τι αφορά τη μη εφαρμογή, γιατί αυτό είναι πολύ σημαντικό και γίνονται πάρα πολλές ε, ατασταλίες και ανακρίβειες. Ε, γιατί έχουμε την εντύπωση πολλές φορές ότι κάποιος με ένα άτομο με αναπηρία είναι ένα άτομο το οποίο ούτως ή άλλως έχει τα προβλήματά του και δεν χρειάζεται να το φροντίσουμε. Αυτό είναι απαράδεκτο. Ξεκάθαρα χρονοδιαγράμματα, ποινικέ ε, κυρώσεις αν δεν γίνεται σωστή εφαρμογή και τρίτον σαφής διαχωρισμός για τον τομέα εφαρμογής και ισχύω. Και αυτό θα πρέπει με ακρίβεια να ρυθμίζεται. Καταλαβαίνω τι λέει ο συνάδελφος Evans. Αν πρόκειται για βοηθήματα όπου χρειάζεται κανεί πραγματικά σημαντική βοήθεια από κάποιον άνδρα, από κάποια γυναίκα, είναι προβληματική η κατάσταση. Γιατί το άτομο αυτό ίσως να μην έχει αρκετή δύναμη, να μην έχει κάποιο άτομο να τον συνοδεύσει. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς θα πρέπει να εφαρμοστεί κάτι τέτοιο. Φυσικά θα πρέπει να πετύχουμε αυτό που θέλουν και οι ενώσεις αναπήρων. Θέλουν όσο το δυνατόν πιο ανεξάρτητα να κινούνται και μόνοι τους, χωρίς διαρκώς να πρέπει να παρακαλέσουν για βοήθεια. Και αυτό παρακαλώ να αποτελεί και ένα από τις, μία από τις βασικές αρχές του θέματος αυτού. Αυτή η εξάρτηση, αυτή η ανάγκη να ζητήσει κανείς βοήθεια από κάποιον άλλον, να περιοριστεί όσο το δυνατόν γίνεται αναφορικά με τις τεχνικές προδιαγραφές οι οποίες θα πρέπει να πληρούνται. Αυτό να το ξεκαθαρίσουμε γιατί δεν έχει αναφερθεί με ακρίβεια, με αρκετή ακρίβεια στην έκθεση. Το ότι τα πράγματα είναι λίγο πιο δύσκολα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις το καταλαβαίνω, αλλά μιλάμε για ένα θεμελιώδες δικαίωμα. Δεν υπάρχει οποιαδήποτε δικαιολογία για την κατάργηση αυτού του θεμελιωδούς ε, δικαιωμάτων. Το μόνο που μπορεί να δεχτώ είναι κάποιες ιστορικές, αν θέλετε, στάσεις λεωφορείων, τις οποίες ε, δεν θέλουμε για ιστορικούς και συναισθηματικούς λόγους να αλλάξουμε. Ό,τι όμως συγκαταλέγεται στις μοντέρνες σύγχρονες μεταφορές θα πρέπει να αναδιαμορφωθεί και με τον στόχο να αναπτυχθεί μία μέθοδος, ένα σύστημα προκειμένου να μην υποχρεώνεται κανείς να ζητά βοήθεια για να ανέβει στο λεωφορείο. Μπορεί να επιτραπούν κάποιες εξαιρέσεις για μία μεταβατική περίοδο, αλλά όλα αυτά θα πρέπει να ρυθμίζονται με σαφήνεια, να μετρώνται με σαφήνεια και να υπάρχουν και συγκεκριμένα μέτρα. Ιδάλλως δεν θα το πετύχουμε ποτέ. Γιατί μιλάμε εδώ και 30 χρόνια στην Ευρώπη για την ισότητα των αναπήρων, αλλά δεν έχουμε πετύχει ακόμα αυτό που θα έπρεπε να πετύχουμε. Πρόκειται για μια επένδυση, γιατί πάντα ευχόμαστε και ζητάμε να γίνουν επενδύσεις και αυτό θα ήταν το καλύτερο επενδυτικά προγράμματα για ε, προϊόντα στην αυτοκινητοβιομηχανία, αν υπάρξει για παράδειγμα μετεκπαίδευση των ατόμων αυτών, νομίζω ότι κάτι θα έχουμε πετύχει και για πολλούς είναι πολύ σημαντικό το θέμα αυτό. Για τα μέσα μεταφοράς για ένα άτομο και αυτά τα κλασικά coaches που ανέλαβε, ανέφερε ο κ. Evans θα πρέπει να τα ορίσουμε με ακρίβεια, γιατί ιδάλλως θα έχουμε προβλήματα. Ξέρω ότι θα έχουμε πολλές παρεμβάσεις, γιατί είναι εξαιρετικά δυσάρεστο πάντα να αλλάζουμε συστήματα σε ό,τι αφορά τις ε, μεταφορές, αλλά μιλάμε για θεμελιώδη δικαιώματα πολύ απλά, τα οποία θα πρέπει να εφαρμόζονται. Ο κύριος Γιαζεμπόφσκι, είχα ζητήσει το λόγο εδώ και ώρα, κύριε Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω τον συνάδελφο για την εξαιρετική του έκθεση. Σας παρακαλώ, συνάδελφε Κράμερ, να πω δύο πράγματα προς την ε, συνάδελφο Λίχτενμπεργκερ. Δεν ε, έχει νόημα να απευθύνεται και να εκφωνείτε ωραίες ομιλίες, να υποβάλλετε τροπολογίες. Μιλάτε για θεμελιώδη δικαιώματα, αλλά για προσέξτε λίγο, γιατί κοιτώ και το γερμανικό σύνταγμα και τη χαρτό των ε, δικαιωμάτων. Θα πρόσεχα τι λέω. Φυσικά μπορούμε και να ζητήσουμε να υπάρχει αλλαγή στα συστήματα των λεωφορείων και στις στάσεις, Αλλά ίσως με τον τρόπο αυτό θα καταστρέψετε και τις επιχειρήσεις θα πρέπει λοιπόν να προσέχουμε τι αναφέρουμε ως θεμελιώτες δικαίωμα. Επίσης, να πω το εξή. Όλοι θέλουμε να κάνουμε κάτι για τους ανάπηρους, όπως λέει και το κεφάλαιο 3, αλλά αυτά τα δικαιώματα επιβατών δεν ε, ισχύουν μόνο για τους αναπήρους, αλλά για όλους τους πολίτες. Γι' αυτό λοιπόν το κεφάλαιο 4 αναφέρει τα δικαιώματα όλων και μιλάμε ποια είναι η ευθύνη για παράδειγμα σε περίπτωση μεγάλης καθυστέρησης και αυτό ανέφερε και ο συνάδελφος ε, Evans που μίλησε για το coaches, για τα πούλμαν και σε ό,τι αφορά τις μεταφορές αυτές ή τις ε, αεροπορικές μεταφορές αν υπάρχει κάποιος εύλογος λόγος καθυστέρησης θα πρέπει να προστατεύεται ο επιβάτης. Μιλάμε όμως για τον κανονικό επιβάτη. Αυτόν έχουμε καταρχάς υπόψη μας. Έχω τρεις τροπολογίες. Για το κεφάλαιο 8, παράγραφος 1. Νομίζω ότι θα πρέπει να είμαστε λίγο πιο ακριβείς. Μιλάμε για τις πληρωμές σε περίπτωση θανάτου ή ατυχήματος ή οποιαδήποτε βλάβης της σωματικής και πνευματικής υγείας. Καμιά φορά σοκάρουμε από το πώς οδηγούν οι οδηγοί λεωφορείων, αλλά δεν νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει τέτοια νομική ευθύνη. Σε σωματική βλάβη ή σε περίπτωση θανάτου, εντάξει. Γιατί θεωρώ ότι καμιά φορά οι οδηγοί λεωφορείων είναι πραγματικά διδραγμένα άτομα, αλλά δεν ξέρω. Και επίσης αυτή η ρύθμιση, η ρήτρα για την ευθύνη είναι σωστή, είναι πολύ αυστηρή, αλλά μου λείπει και μία δεύτερη παράγραφος, όπου θα, μάλλον, που θα αναφέρεται ότι σε περιπτώσεις ανώτερης βίας απαλλάσσεται η επιχείρηση. Γιατί υπάρχουν άλλωστε και ανάλογες αποφάσεις του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σε περίπτωση ανώτερης βίας. Θα πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία. Θέλουμε να προστατεύσουμε τα δικαιώματα των επιβατών, αλλά θα πρέπει να προστατεύσουμε και τα δικαιώματα των ε, επιχειρήσεων. Αν έχει πέσει ένα δέντρο δηλαδή και δεν μπορεί η επιχείρηση να παρέχει τις υπηρεσίες της, δεν μπορούμε να τη θεωρήσουμε υπεύθυνη. Νομίζω ότι αυτό είναι πασιφανές. Και στην παράγραφο 22 για τις περαιτέρω αξιώσεις, νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρξει μία αναδιατύπωση, όπως και στον κανονισμό, για να μην υπάρχουν διαφορετικές διατυπώσεις. Αλλά νομίζω ότι αυτά είναι μάλλον λεπτομέρειες, θα τις υποβάλω συνάδελφε και κατά τα άλλα θεωρώ ότι είναι εξαιρετική η έκθεση και ανυπομονώ να δω και τι θα ακούσουμε και στη μελλοντική συζήτηση. Also äh, Ο κύριος Κράμερ, όταν μιλάμε για δικαιοσύνη, ε, 30% των οδηγών στην ε, κίνηση στις δυνατικές μεταφορές ε, είναι ανάπηροι και αυτό δεν αφορά μόνο τα άτομα σε αναπηρικά καροτσάκια, αφορά και ηλικιωμένους, ε, αφορά πατέρες με μικρά παιδιά, άτομα τα οποία κυκλοφορούν ε, ένα μήνα με γύψο στο πόδι και υπάρχει μάλιστα ένας σχετικός καθηγητής ε, πανεπιστημίου ο οποίος έχει συστήσει στους φοιτητές του να κυκλοφορήσουν δύο εβδομάδες με γύψο στο πόδι στη Στουγκάρντι για να δουν τι ακριβώς σημαίνει αναπηρία. Και ξέρουμε ότι περίπου το 20% των οικοκυριών δεν έχουν αυτοκίνητο. Δηλαδή όσο πιο πολύ ε, γερνάει ο άνθρωπος, επίσης τόσο λιγότερο, τόσο πιο πολύ εξαρτάται από τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Χρειαζόμαστε λοιπόν να το λάβουν αυτό υπόψη όλοι οι θεσμοί. Και φυσικά και τα οχήματα τα οποία μετακινούνται στον δρόμο. Αν το συγκρίνουμε αυτό με την υπόλοιπη Ευρώπη, διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν διαφορές. Αλλά είχα πάει και στις ε, Ηνωμένες Πολιτείες και σε κάθε λεωφορείο, μα σε κάθε λεωφορείο υπάρχει δυνατότητα να μπει κανείς με αναπηρικό καρατσάκι. Παίρνει λίγη ώρα και ο οδηγός βοηθάει, δεν είναι και το καροσάκι. Σε κάθε λεωφορείο σε κάθε λεωφορείο και πρέπει να σας πω ότι καμία φορά δεν διαμαρτυρήθηκε ούτε ένας επιβάτης γιατί πολλές φορές είδα να μπαίνει ένα παιδικό καρατσάκι και γιατί ε, υπάρχει αλληλεγγύη. Ρώτησα λοιπόν γιατί αυτό ισχύει στην Αμερική ιδιαίτερα γιατί υπάρχει ε, ομοσπονδιακός νόμος και αυτό μετά τον πόλεμο γιατί βρέθηκε η Αμερική με πολλούς ανάπηρους πολέμου και ξαφνικά λοιπόν προβλέφθηκε αυτή η δυνατότητα για τους ανάπηρους πολέμου και κατέστη αυτό υποχρεωτικό για όλα τα λεωφορεία. Άλλα λεωφορεία που δεν έχουν τέτοια δυνατότητα δεν παράγονται καν. Αποτελεί πρότυπο αυτό. Αν αυτό λοιπόν ήταν δυνατόν να γίνει για τους ανάπηρους του πολέμου του Βιετνάμ, γιατί δεν μπορεί να γίνει αυτό για μια κοινωνία των πολιτών που δεν έχει αντιμετωπίσει και το έξοδο του πολέμου, τις δαπάνες του πολέμου. Θα πρέπει να επιβάλλουμε πιο αυστηρέ προδιαγραφέ. Αυτά που συζητάμε, αυτό λοιπόν που μπόρεσαν και πετύχαν οι Ηνωμένε Πολιτείε, θα έπρεπε να μπορεί να το, ε, μπορεί να το πετύχει και η Ευρώπη. Γι' αυτό λοιπόν θεωρώ ότι η αποδοχή είναι τεράστια. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε, να δημιουργήσουμε το σχετικό πλαίσιο και γι' αυτό πρέπει να το δημιουργήσουμε. Κύριε Γέγκλε, ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και μετά από αυτά που είπατε, κύριε Κράμερ, θα ήθελα να αναφερθώ σε αυτά που είπε και ο Βρετανός συνάδελφος. Νομίζω ότι όλα τα μέσα θα πρέπει να εξυπηρετούν τον σκοπό μας. Είναι σωστή η προσέγγιση αυτή, αλλά η έκθεση αναφέρει και το πρόβλημα των καθυστερήσεων. Και αν το συνδυάσουμε αυτό θα πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί, δεν θα πρέπει να δημιουργούμε προσδοκίες οι οποίες ενδεχομένως να μην πραγματοποιηθούν. Αν πάω από την Νότια Γερμανία στη Μεγάλη Βρετανία, για να αναφερθώ και στο θέμα της καθυστέρησης, στο νότο της Γερμανίας ε, το δίκτυο των μεταφορών είναι αρκετά εκτεταμένο, να το πούμε έτσι. Μάλλον ε, μπορεί να αναπτυχθεί και παραπάνω. Τι καθυστερήσεις αντιμετωπίζω, για παράδειγμα στο Λουξεμβούργο ή στο Βέλγιο, όταν λαμβάνω επιβάτες. Η πρώτη στάση φταίει ή η δεύτερη στο Βέλγιο, στο Λουξεμβούργο, για την οποία δεν ευθύνεται η επιχείρηση του λεωφορείου Και η συμφόρηση στους γερμανικούς δρόμους, αυτό θα πρέπει να το σκεφτούμε και καταλαβαίνω την κατάσταση που πλήττει τους αναπήρους. Μιλήσατε για 30%, η Κομισιόν αναφέρει 40%. Τι κάνουμε λοιπόν. Νομίζω ότι θα πρέπει να βρούμε τα απαραίτητα μέσα για να παραδώσουμε μια καλή έκθεση η οποία ούτε υπερβολικές προσδοκίες θα δημιουργεί και επανέρχομαι και πάλι σε αυτό που είπε ο Βρετανός συνάδελφος γιατί προσανατολιζόμαστε τη συνδυασμό διαφόρων τρόπων μεταφοράς, να κοιτάξουμε τα στοιχεία αυτά τα οποία θα πρέπει να λειτουργούν σε διεθνές, σε διεθνές επίπεδο και κατά τα άλλα να τηρήσουμε και ε, τη σχετική νομοθεσία. Ευχαριστώ. Evans. Ο κύριος Evans. Να επανέλθω σε ένα-δυο σημεία. Η κυρία Γέγκλη έκανε μια πολύ σημαντική παρατήρηση για αποζημιώσεις ε, σε μακροχρόνια ε, ταξίδια και καθυστερήσεις. Αυτό που θα πρέπει να κάνουμε είναι ή να βρούμε την κατάλληλη δια, ε, ή να διευκρινίσουμε σαφώς ότι όταν οι καθυστερήσεις δεν οφείλονται σε κυκλοφοριακή κίνηση, αλλά είναι ευθύνη είτε του λοφορίου είτε της εταιρεία ε, των λεωφορείων, ε, να μην υπάρχει μια μικρή, ένα μικρό παραθυράκι που να μπορούν να πούν ότι «Α, είχε πολύ κίνηση στο Λουξεμβούργο και γι' αυτό καθυστερήσαμε». Ε, ορισμένοι από αυτούς ε, έχουν καταφέρει πάρα πολύ καλά να λένε ότι α, ε, δεν ισχύει ο κανονισμός ε, στις αεροπορικές εταιρείες γιατί υπήρχε άλλη συγκεκριμένη καθυστέρηση και δεν φταίμε εμείς, επομένως δεν ισχύει ο κανονισμός για τις αποζημιώσεις. Πρέπει λοιπόν να σκεφτούμε την κατάλληλη διατύπωση προκειμένου να μην δοθεί κανένα παραθυράκι διεξόδου για να λέμε ότι είχαμε καθυστέρηση, είχε κίνηση στο δρόμο και αυτό καθυστέρησε το πούλμαν ή να πιέσουμε τον ίδιο τον οδηγό, διότι αν η καθυστέρηση του λεωφορείου είναι μεγαλύτερη από δύο ώρες, ε, σημαίνει ότι ο οδηγός θα πιεστεί πάρα πολύ για να κάνει ένα ε, ταξίδι το οποίο θα χρειαζόταν δύο ώρες να το κάνει ε, και θα το κάνει σε μια μισή ώρα για να μην χρειαστεί να πληρώσει την υποζημίωση. Αυτό είναι κάτι ακόμα που πρέπει να λάβουμε υπόψη. Να σταθώ και σε κάτι που είπε ο κύριος Γερζεμπόφσκι. Νομίζω ότι το σημείο ακριβώς όπως το είπατε. Είπατε ότι δεν μιλάμε μόνο για τα δικαιώματα των αναπήρων, μιλάμε και για τους καθημερινούς πολίτες. Εγώ θα ήθελα να πω ότι οι ανάπηροι είναι καθημερινοί πολίτες, είναι συνηθισμένοι άνθρωποι και αυτούς αφορά η οδηγία. <laughs> Ευχαριστώ πολύ όλους τους συναδέλφους για την ε, Κομισιόν τώρα, η εκπρόσωπος. Παρακαλώ. Uh, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον εισηγητή για την πολύ καλή αυτή έκθεση και την πολύ καλή συνεργασία. Θα ήθελα να σας επιθυμίσω τους βασικούς στόχους Ευρωπαϊκής Επιτροπής εναρμόνιση ουσιαστικά των δικαιωμάτων των επιβατών για όλα τα μέσα μεταφοράς. Αυτό αποτελεί πλέον πάγια τακτική της ε, ευρωπαϊκής πολιτικής μεταφοράς ήδη από τη Λευκή Βίβλο του 2001. Προτείναμε μια νέα προσέγγιση το 2005 με ειδική ανακοίνωση Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα δικαιώματα των επιβατών και στη συνέχεια υπήρξε πολύ σημαντική δέσμευση Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην ενδιάμεση αναθεώρηση του 2006 για να καταφέρουμε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα στη μεταφορά επιβατών σε όλα τα μέσα μεταφοράς. Πιστεύουμε ότι οι επιβάτες θα πρέπει να αναγνωρίζουν τα δικαιώματά τους, αυτά να είναι ευνόητα και να μπορούν εύκολα να εφαρμοστούν. Προσπαθούμε επίσης να έχουμε νομοθεσία εξειδικευμένη για κάθε τομέα και να έχουμε και έξι κοινέ αρχές. Η πρώτη είναι ότι δεν θα πρέπει να υπάρχει εμπορική διακριτική μεταχείριση μεταξύ των επιβατών όσον αφορά τις τιμές ή τις συνθήκες μεταφοράς ταξιδιού. Δεύτερον, οι επιβάτες θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το ταξίδι. Τρίτον, οι επιβάτες θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε αποζημίωση σε περίπτωση ατυχήματος και θα πρέπει να εναρμονιστούν τα συστήματα ευθύνης για όλες τις επιχειρήσεις μεταφορών. Τέταρτον, τα άτομα με αναπηρίες και τα άτομα με μειωμένη κινητικότητα θα πρέπει να έχουν εγγυημένη πρόσβαση στις υπηρεσίες μεταφορών κατά τον ίδιο τρόπο, με τον ίδιο τρόπο όπως ισχύει ουσιαστικά για όλους τους επιβάτες. Πέμπτον, σε περίπτωση αλυσιδωτών ταξιδιών θα πρέπει οι ε, επιβάτες σε περίπτωση με συγχωρείτε διακοπής του ταξιδιού θα πρέπει οι επιβάτες να έχουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και θα πρέπει επίσης να δίνεται και η απαραίτητη αποζημίωση. Εφόσον αυτό χρειαστεί βέβαια. Και τέλος θα πρέπει να υπάρχουν κατάλληλες διαδικασίες εξοδικαστικής διευθέτησης διαφορών που να προκύψουν μεταξύ επιχειρήσεων και επιβατών. Καταλαβαίνετε ότι μολονότι έχουμε τις έξι αυτές κοινέ αρχές, δεν σημαίνει ότι θα έχουμε κοινή και ίδια αντιμετώπιση όλων των τομέων. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας τις ιδιαιτερότητες κάθε τομέα, για παράδειγμα στον ε, τομέα της ε, αεροναυτιλίας. Αυτό που μας ενδιαφέρε περισσότερο ήταν ε, το δικαίωμα μιας αεροπορικής εταιρείας να μην επιτρέψει την επιβάτη να ταξιδέψει. Στον οδικό τομέα έχουμε άλλες άλλα στοιχεία τα οποία μας απασχολούν και πιο συγκεκριμένα το ζήτημα της αποζημίωσης σε περίπτωση καθυστέρησης. Μέσω της εφαρμογής των πρώτερων κανονισμών όσον αφορά την αεροναυτιλία και όσον αφορά επίσης ε, την εφαρμογή του κανονισμού εκείνου που είχε να κάνει με την ε, αεροναυτιλία και τις δρομικές μεταφορές έχουμε καταφέρει να αποκομίσουμε την απαραίτητη εμπειρία που θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε και σε αυτή την πρόταση κανονισμού. Βέβαια, δεν έχουμε ακόμα ασχοληθεί δεόντως με το ζήτημα της υποδομής και το ζήτημα της ε, προσβασιμότητας των ε, οχημάτων. Και αυτό προσπαθήσαμε να το κάνουμε τις προτάσεις που υποβάλαμε το Δεκέμβριο. Προσπαθούμε επίσης να θεσπίσουμε κοινού κανόνες όσον αφορά την προστασία των καταναλωτών ε, βάσει του τόπου που παρέχεται η υπηρεσία ή βάσει του τρόπου μεταφοράς. Θέλουμε να έχουμε πλέον μια κοινή πολιτική προστασία των καταναλωτών, η οποία να μπορεί να εφαρμοστεί ομοιόμορφα σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ και την κυρία Ούτμαν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Άκουσα με ιδιαίτερη προσοχή. Σημείωσα και πάρα πολλά πράγματα ε, στα όσα είπαν οι συνάδελφοι. Θεωρώ ότι στο σύνολό τους είναι πάρα πολύ ισορροπημένα τα σχόλια και ιδιαίτερα ε, χρήσιμα. Συμφωνώ με τον ε, κύριο Εύανς ότι θα πρέπει να λάβουμε υπόψη πολύ καλά τον γενικό στόχο που είναι να διασφαλίσουμε ότι θα έχουμε κοινά δικαιώματα για όλους τους επιβάτες, ε, ακόμα και τους... Ε, τα άτομα με αναπηρία γιατί ούτως ή άλλως και αυτοί είναι επιβάτες όπως όλοι, τους, όπως όλοι οι άλλοι και αυτό θα πρέπει να ισχύει για όλες τις χώρες και για όλα τα μέσα μεταφοράς λαμβάνοντας υπόψη λογικά την ιδιαιτερότητα ε, της κάθε πτυχής ε, όσον αφορά σε θέματα διαχείρισης. Να ευχαριστήσω και τον κύριο Ρη, συμφώνησες για όλα σχεδόν, όσον αφορά στην τροπολογία 10 θα εμβαθύνουμε το δίχως άλλο στα θέματα τα οποία ανέφερες. Κυρία Λίχτεμπεργκ, εσείς εκφράσατε όχι ακριβώς τη διαφωνία σας, αλλά μία αίσθηση συνένεσης. Ε, είναι πολύ σημαντική αυτή η επισήμανση που κάνετε. Το χρονοδιάγραμμα που έχετε προτείνει, όπως σας είπα ήδη, είναι το ενδιάμεσο χρονοδιάμενα, δηλαδή ε, δύο χρόνια για την εφαρμογή, διότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητούσε ένα χρόνο και δεν λαμβάνει υπόψη της τις πολυάριθμες καθυστερήσεις που είχατε πει και όπως επίσης αυτό το οποίο που πρότειναν οι μεταφορείς οι οποίοι ζητούσαν τρία χρόνια. Τώρα, όσον αφορά στην παρέμβαση του φίλου και συναδέλφου Γερζεμπόσκη, συμμερίζομαι τα όσα είπε ε, με αφηρημένο τρόπο. Δηλαδή, με τα όσα είπατε, εάν αναφέρεστε στην περίπτωση της Γερμανίας, διότι μελέτησα μαζί σας και τους εκπροσώπους των ασφαλιστικών εταιριών ε, τα προβλήματα ανωτέρας βίας, τα οποία είναι τέλεια από νομικής πλευράς. Το δικό μου το πρόβλημα, ως Ιταλός, και λαμβάνοντας υπόψη και υπάρχει και μια συγκεκριμένη νοοτροπία που κάποιες χώρες που διαφέρουν από τη Γερμανία που είναι τόσο αυστηρή και ακριβής ακόμα και στην ομολογία της ε, μπορεί να αναπτύξουν και να αντιμετωπίσουν, ε, θεωρούμε ανωτέρα βία οποιαδήποτε περίπτωση ε, μπορεί με χαλαρό τρόπο να θεωρηθεί κάτι τέτοιο. Δηλαδή δεν θα ήθελα από αυτή την εξαιρετική έννοια της ανωτέρας βίας να διευρύνουμε το πεδίο εφαρμογή σε οποιαδήποτε άλλη δυνατότητα διότι αυτό θα παρενέβαινε τις γενικές αρχές τις οποίες πρέπει να τηρήσουμε. Πολύ σωστές οι σκέψεις του συναδέλφου Κράμερ ως προς την συγκεκριμένη μέρημνα για τους αναπήρους, ε, ένα από τους βασικούς στόχους, όπως υπενθύμησε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτού του κανονισμού, είναι να υπάρχουν πανομοιότυπα δικαιώματα για όλους τους Ευρωπαίους πολίτες σε οποιαδήποτε κατάσταση και αν βρίσκονται, σε οποιαδήποτε προσωπική κατάσταση μειωμένης ε, προσωρινής ή σταθερής κινητικότητας και για οποιοδήποτε μεταφερικό μέσο χρησιμοποιούν. Γι' αυτό ακριβώς και ο δικός μας ο κανονισμός ε, συνδέεται με τους υπόλοιπους ε, και με το σύνολο της νομοθεσίας που αφορά τις ε, θαλάσσιες, ποτάμιες, εναέριες, σιδηροδρομικές μεταφορές και οποιαδήποτε άλλη. Τώρα, για κάποια άλλα σημεία πιο διεξοδικά Νομίζω ότι θα μπορούσαμε να συζητήσουμε περαιτέρω στους διαλόγους που θα κάνουμε. Σας επαναλαμβάνω ότι από τις επόμενες κιόλας ώρες θα συναντήσω τους κοιόδης συζητητές από όλε τις ε, πολιτικές ομάδες, αλλά η εντύπωση που αποκόμισα από αυτή την τόσο ε, ενδιαφέρουσα και εις βάθος συζήτηση, παρά το γεγονός ότι συζητήσαμε για λίγο χρονικό διάστημα, είναι ότι σε γενικές γραμμές είμαστε όλοι θετικά διακείμενοι ως προς την ε, τοποθέτησή μου για, την, ε, ε, για το κατά πόσο θα πρέπει να προσπαθήσουμε να επιτύχουμε κάποιους στόχους και θεωρώ ότι ξεκινούμε από τις βέλτιστες συνθήκες και βούλησης και συνεργασίες προκειμένου να φτάσουμε σε ένα καλό αποτέλεσμα εντός των στενών προθεσμιών που θέλουμε να επιτύχουμε, δηλαδή έγκριση στην Ολομέλεια μέχρι τον Απρίλιο. Σας ευχαριστώ και για άλλη μια φορά για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε τον κύριο Αλμπερτίνη. Τροπολογίες, προθεσμία μέχρι τις 2 Μαρτίου ή αλλιώς δεν έχετε άλλο χρόνο. Να περάσουμε τώρα στο σημείο υπαριθμών 28, δικαιώματα των επιβατών. Α, συγγνώμη, Μάρτιο, 2 ε, Μαρτίου 12. Ε, δικαιώματα των επιβατών θαλάσσιων και εσωτερικών πλωτών μεταφορών. Ο κύριος Τεσενέ έχει το λόγο. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η συζήτηση που μόλις ε, κάναμε θα μας βοηθήσει να, να καταλάβουμε περισσότερο την έκθεση που θέλω εγώ με τη σειρά μου να σας παρουσιάσω. Επίσης, η παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μας υπενθύμησε τις έξι βασικές αρχές Ευρωπαϊκής Επιτροπής που διέπουν και τη δική μου την έκθεση. Όσον αφορά πιο συγκεκριμένα τα δικαιώματα των επιβατών θαλάσσων και εσωτερικών πλωτών μεταφορών, θα ήθελα να σας πω ότι ε, επικεντρώθηκα περισσότερο στα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία και μειωμένη κινητικότητα, προκειμένου να καταφέρουμε να συντοπίσουμε καλύτερα τα δικαιώματά τους και να αποφύγουμε τη δημιουργία εξαιρέσεων που θα δίνουν τη δυνατότητα σε επιχειρήσεις να μην προστατεύουν τους ε, πολίτες αυτούς. Όπως ε, για παράδειγμα η δυνατότητα μιας επιχείρησης να αρνηθεί την επιβίβαση σε έναν άνθρωπο με αναπηρία σε ένα πλοίο. Επίσης, θέλουμε επίσης να υπάρχουν συγκεκριμένε διατάξεις όσον αφορά την αρρωγή προς τα άτομα αυτά με αναπηρία και μειωμένη κινητικότητα και να περιγράφονται συγκεκριμένα οι ευθύνες που φέρει προς τα άτομα αυτά μια επιχείρηση θαλασσίων μεταφορών. Επίσης, θέλουμε να καλύψουμε και τις κουραζιέρες στην έκθεση αυτή και θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας διατάξεις που ήδη ισχύουν στην υφιστάμενη οδηγία του 1991 η οποία επικεντρώνεται στις κουραζιέρες προσπαθήσαμε να πετύχουμε την κατάλληλη ισορροπία, αν θέλετε, ανάμεσα στον κανονισμό αυτό και την οδηγία του 1991. Τώρα, περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά την αρρωγή προς τα άτομα με αναπηρία και μειωμένη κινητικότητα όταν βρίσκονται στο λιμένα. Στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής βλέπουμε περισσότερο τις ευθύνες που φέρει ο μεταφορέας. Ευθύνες όμως φέρουν και οι ίδιοι λιμένες. Επομένως θα πρέπει να υπάρχει εδώ η απαραίτητη υποδομή προκειμένου να παρέχεται κατάλληλη βοήθεια στα άτομα με μειωμένη κινητικότητα. Υπέβαλα λοιπόν ως προς αυτό κάποιες τροπολογίες προκειμένου να γίνει μια καλύτερη συζήτηση και μια καλύτερη εναρμόνιση των ευθυνών που φέρουν από τη μια η φορείς διαχείριση νοσλημένα και από την άλλη η μεταφορείς. Επίσης αναφέρομαι στο ρόλο των εθνικών φορέων που είναι ταγμένοι να εξασφαλίζουν την εφαρμογή του μελλοντικού κανονισμού. Ο ρόλος τους ενισχύεται και διασαφηνίζεται στο κείμενο αναφέρονται διάφοροι οργανισμοί, νομίζω θα ήταν καλύτερο να έχουμε έναν κοινό οργανισμό για να πετύχουμε την κατάλληλη εναρμόνιση. Οι ε, οργανισμοί αυτοί θα κληθούν να φέρουν μια μεγαλύτερη ευθύνη, κυρίως όσον αφορά την ε, μη διακριτική πρόσβαση στις μεταφορές θαλασσίων και εσωτερικών πρωτών μεταφορών στα άτομα αναπηρία και μειωμένη κινητικότητα. Επίσης θεωρώ ότι οι οργανισμοί αυτοί θα πρέπει να λειτουργούν ανεξάρτητα από τα εμπορικά συμφέροντα. Επιβάλλεται λοιπόν η εξαρτησία τους και πρέπει αυτή να εξασφαλιστεί. Τέλος, όσον αφορά τις μεταφορές, προσπάθησε να δώσω μεγαλύτερη ακρίβεια στους ορισμούς σχετικά με τις συμβάσεις μεταφοράς, τους πολιτές εισιτηρίων και τους ε, ταξιδιωτικούς πράκτορες. Θέλουμε να γνωρίσουμε εδώ πέρα ποιος είναι, ποιος τι ακριβώς γίνεται, ποιος είναι υπεύθυνος για τις κρατήσεις και για τις μεταφορές. Επίσης, ε, κάνουν έκκληση για μια διοικητική απλούστευση εφόσον αναφερόμαστε εδώ πέρα σε κείμενα τα οποία έχουν να κάνουν και με τις αεροπορικές μεταφορές. Πολλές φορές μέσω του κειμένου αυτού θα αναγκάζαμε κάποιες επιχειρήσεις να έχουν δύο συστήματα λογιστικά, πράγμα το οποίο γίνεται αυτή τη στιγμή για τις αεροπορικές εταιρείες, αλλά θα ήταν πιστεύω ιδιαίτερα δύσκολο για τις μικρές επιχειρήσεις θαλασσίων και εσωτερικών πλωτών μεταφορών. Επίσης, όσον αφορά πιο συγκεκριμένα τις ποτάμιες μεταφορές, πιστεύω ότι θα πρέπει να ενσωματωθούν πλήρως στο κείμενο εφόσον βλέπουμε ότι όλο και περισσότεροι μεταφορείς ε, ποταμίων ε, μεταφορών εμπλέκονται πλέον και στις αστικές μεταφορές, πολλές φορές ε, μέσα στα όρια μιας πόλης και εφόσον γίνονται αναφορές και στις κρουαζιέρες μέσα στο κείμενο αυτό. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να ενσωματωθούν και αυτές οι αστικές πλωτές μεταφορές. Αυτά όσον αφορά τις αρχικές παρατηρήσεις ε, που ήθελα να κάνω για την έκθεση αυτή και επαφίομαι βέβαια και στη βοήθεια των συναδέλφων. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Ζεμπόφσκι, ευχαριστώ πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, να πω στον ε, Πρωτάρη εισηγητή ότι είναι εξαιρετική η έκθεσή του, σας συγχαίρω. Σας συγχαίρω εκ μέρου τη ομάδα μου. Για το τελευταίο αυτό θέμα νομίζω ότι θα πρέπει να επικεντρωθούμε στο μέσο και παρά το γεγονό ότι το πλοίο κινείται όπω το λεωφορείο εξακολουθεί να είναι πλοίο. Δεν μπορούμε να τα συγχαίουμε αυτά. Δεν είναι το πλοίο τετραόροφο Λεωφορείο, να μην τα συγχαίουμε αυτά. Έχω κανένα δύο ερωτήσει τις οποίες θέλω να σας θέσω και να υποβάλω και τροπολογίες. Αυτό που ανέφερα και για την έκθεση Λαβερτίνη, το θέμα είναι το θέμα της αποζημίωσης για τις καθυστερήσεις. Μπορούμε να το επιβάλλουμε στις επιχειρήσεις μόνο εάν ευθύνονται όντως για την καθυστέρηση αυτή και μπορούσαν να την αποτρέψουν. Και ίσως εδώ στις ε, ναυτιλιακές μεταφορές θα πρέπει να εισαχθεί και ένας ειδικό όρος στον τομέα της ε, Βορείου Ευρώπης, στη Βαλτική. Αν ε, τίθεται θέμα πάγου για παράδειγμα, δεν μπορεί να ταξιδέψει το πλοίο και πρόκειται για ένα παράδειγμα για το οποίο δεν είναι υπεύθυνη η επιχείρηση. Έχουμε για παράδειγμα και στα γερμανικά νησιά σημεία με πολύ μεγάλο βάθος, πυθμένα, που μπορεί να αποτελέσουν πρόβλημα σε περίπτωση που υπάρχει παλήρια για τα πλοία. Πρόκειται για μια συνήθιστη κατάσταση για την οποία δεν ευθύνεται η επιχείρηση. Αυτό θα πρέπει να το διευκρινίσουμε. Μια άλλη παρατηρήση τώρα. Ε, μια πρακτική ερώτηση μάλλον. Στο άρθρο 13 πρόκειται αναφέρονται οι υποχρεώσεις ε, ανακοίνωσης, ενημέρωσης. Μου φαίνεται ότι είναι πολύ πολύπλοκη η κατάσταση. Θα πρέπει δηλαδή να αναφέρεται, υπάρχει υποχρέωση αναφοράς σχετικά με ποια μέσα είναι απαραίτητα και χρειάζονται. Δηλαδή ο ένας υπεργολάβος θα πρέπει να ενημερώσει τον άλλο υπεργολάβο για να ενημερώσει τον τρίτον υπεργολάβο. Τελικά κανείς δεν θα αισθάνεται υπεύθυνο. Αλλά νομίζω ότι θα φτάσουμε και σε αυτό, θα το κοιτάξουμε με την ησυχία μας. Θεωρώ ότι είναι εξαιρετική η έκθεση. Και μόνο αυτά τα θέματα έχω. Τι γίνεται για τις, με τις εξαιρετικές ε, αυτές περιπτώσεις, για παράδειγμα σε περίπτωση παλήριας ή παγετώνα. Κυρία Λίχτενμπέργκερ, ευχαριστώ για τα δικαιώματα των επιβατών στη θάλασσα. Νομίζω ότι έχουμε να διορθώσουμε πάρα πολλά και σε ό,τι αφορά τα άτομα με αναπηρία και με ειδικές κινητικές ανάγκες. Μία ερώτηση να σας θέσω. Έχουμε παρόμοια προβλήματα όπως και στους αερολιμένες και με τις αεροπορικές εταιρείες. Ωστόσο, δεν μου φαίνεται ότι είναι συνεκτική η έκθεση σε ό,τι αφορά του ποιος έχει την ευθύνη τελικά, προκειμένου και οι διεπαφές να λειτουργούν μεταξύ του διαχειριστή και του λιμένα. Ο λιμένας, για παράδειγμα, πρέπει να φροντίζει προκειμένου να υπάρχει πρόσβαση σε κάποια πράγματα, αλλά όπου χρειάζεται βοήθεια, ποιος το ρυθμίζει αυτό. Ποιο έχει την ευθύνη προκειμένου τελικά να λειτουργεί σωστά η μεταφορά, γιατί είχαμε το πρόβλημα αυτό και με τις ε, φτηνέ αεροπορικές εταιρείε, οι οποίες ε, έπρεπε να ξαναρυθμίσουν τα του handling στην αερολιμένα. Αυτά θα πρέπει να τα κοιτάξουμε με προσοχή για να δούμε πώς μπορούμε με τον καλύτερο τρόπο να τα ρυθμίσουμε δεν είναι αρκετά ακριβή η έκθεση από αυτή την πτυχή. Θα πρέπει να κοιτάξουμε ίσως ποια θα πρέπει να είναι η ιδανική ρύθμιση για να υπάρχει συνέπεια και συνοχή. Δεύτερο θέμα. Φυσικά υπάρχει και ο παγιτόνας, υπάρχουν και ειδικέ συνθήκες. Αλλά να αποφύγουμε, να αποφύγουμε να αναφέρουμε ως επιχείρημα για την καθυστέρηση ότι είχαμε αντίθετο άνεμο, για παράδειγμα. Γιατί δυστυχώς με τα αεροπλάνα έχουμε δει ότι γίνονται για παράδειγμα υπάρχουν τεχνικές βλάβες όταν δεν είναι πολύ οι επιβάτες στο αεροπλάνο. Αυτά, αυτές οι ρυθμίσεις οι εξαίρεσεις την χάνουν κατάχρησης πολύ συχνά. Για να υπεκφύγει ο μεταφορέας των ευθυνών του. Αυτά λοιπόν θα πρέπει να τα αποφύγουμε. Γιατί πραγματικά αυτό οδηγεί σε αγανάκτηση. Και το είπε και η κυρία Γέγκλε. Ο επιβάτης και δικαίω έχει την προσδοκία ότι μπορεί να χρησιμοποιήσει ένα εναλλακτικό μέτρο. Και στην περίπτωση αυτή εμφανίζεται τεχνική, τεχνικό πρόβλημα. Ε, ο επιβάτης πώς θα βγει και θα πει ότι δεν υπήρχε τεχνικό πρόβλημα ή μάλλον δεν υπήρχε τεχνικό πρόβλημα. Υπό κανονικές συνθήκες, αν δεν υποστεί κανείς ε, μεγάλη ζημία λόγω της καθυστέρησης, ε, δεν προβαίνει και σε δικαστική δίωξη. Θα πρέπει να προβλέπετε λοιπόν μια σαφής διαδικασία, να μιλάμε πραγματικά για εξαιρετικές συνθήκες. Ίσως θα μπορούσαμε να το λύσουμε αυτό μέσω της υποχρέωσης ε, παροχής αποδείξεων για να αυξηθεί η πίεση στις επιχειρήσεις σε περίπτωση, για παράδειγμα, να μην εμφανίζονται περιστατικά τεχνικών βλαβών όταν ε, είναι λίγοι επιβάτες. Νομίζω ότι αυτό το έχουμε δει πάρα πολλές φορές στο παρελθόν και σε κάποιες ε, περιπτώσεις κρεμή και απόφαση του δικαστηρίου. Ίσως λοιπόν θα έπρεπε να το αποφύγουμε αυτό ευθύς εξ αρχής με την έκθεση αυτή και φυσικά, φυσικά υπάρχουν ιδιαίτερε συνθήκες. Και στις θαλάσσιες μεταφορές, αλλά θα πρέπει, όπως σας είπα, να υπάρχουν καλές και σωστές διατυπώσεις. Να ευχαριστήσω τον εισηγητή που θίγει το θέμα των ε, σκύλων βοήθειας, το οποίο είναι για πολλούς ανάπηρους σημαντικό και ίσως αυτό θα έπρεπε να αποτελέσει μια ιδέα για να το αναφέρουμε και σε ό,τι αφορά τις μεταφορές με λεωφορεία και πούλμαν, γιατί Συχνά υπάρχουν προβλήματα στις ε, μεγάλες αποστάσεις, ε, λιγότερο στις αστικές μεταφορές, αλλά στις μεγάλες αποστάσεις ναι, ίσως θα ήταν σωστό αυτό να συμπεριληφθεί και αυτό. Και εμένα μου αρέσει όμως η έκθεση. Και αν διευκρινίσουμε αυτά τα θέματα που ανέφερα, για να μην ανοίξουμε τους ασκούς ε, του αιώλου και παραθυράκια για διάφορες εξαιρέσεις, νομίζω ότι θα έχουμε πετύχει πολλά θετικά και θα έχουμε πραγματικά συνεκτικές ρυθμίσεις για όλα τα δικαιώματα των επιβατών, για όλους τους τρόπους μεταφορών και κυρίως σε ό,τι αφορά το σύνολο και τους συνδυασμού των μεταφορών. Η κυρία Γέντσεν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ο κύριος Πισκόσκι είναι σκιώδη εισηγητής εξ ονόματο τη ομάδα μα Δεν μπόρεσε να παραστεί σήμερα και γι' αυτό θα ήθελα να πω εξ ονόματο τη ομάδος ότι μπορούμε να δεχτούμε την ε, πλειονότητα του κειμένου, αλλά υπάρχει ένα σημείο στο οποίο έχουμε ένα ερωτηματικό, διότι δεν αντιλαμβανόμεθα τι ακριβώς θέλει ο εισηγητής. Πρόκειται για την ε, τροπολογία υπαριθμών 8 και την τροπολογία 11 λέει ότι ανεξάρτητα με τις διατάξεις του άρθρου 6, οι μεταφορείς μπορούν να αρνηθούν, να εκδώσουν εισιτήρια ή να δεχθούν ε, επί του σκάφους ε, άτομα με περιορισμένη κινητικότητα ή αναπηρία. Αυτό σημαίνει ότι θα μπορούσε κάλλιστα κάποιος να αρνηθεί στον οποιονδήποτε με την οποιαδήποτε είδους αναπηρία την ε, είσοδο επί του πλοίου. Ε, δεν καταλαβαίνω γιατί μπορεί να θέλει κάποιος να κάνει κάτι τέτοιο. Θα ήθελα να μου εξηγήσει λίγο ο εισηγητής από πού προέρχεται αυτή η τροπολογία και να μου εξηγήσει κατά πόσον είναι σωστό και λογικό να αναφέρεται κάτι τέτοιο. Ευχαριστώ. Ο κύριος Σίμψον. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μία πολύ σοβαρή ερώτηση καταρχάς στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διότι δεν είμαι βέβαιος κατά πόσον εντός αυτής της οδηγίας ε, αρχίζουμε να λοξοδρομούμε αναφέρομαι ε, σε διελεύσεις ποταμών και σε τέτοια πράγματα. Δεν ξέρω κατά πόσο λοιπόν περιλαμβάνονται τα ποτάμια. Θα ήθελα να μου διευκρινίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εάν ε, περιλαμβάνονται και αυτές οι ποτάμιες μεταφορές που δεν βγαίνουν στη θάλασσα στην πρόταση. Επίσης, κάτι λιγότερο σοβαρό, δεν ξέρω κατά πόσον ε, οι βάρκες της Βενετίας, οι γόνδολες περιλαμβάνονται, δεν ξέρω αν καλύπτονται και στην έκθεση του κυρίου Αλμπερτίνη ή αν καλύπτονται στην έκθεση του κυρίου Τεσενέ ή μπορεί να καλύπτονται και στα δύο. Ίσως πρέπει να καλύπτονται και από τα δύο οι γόνδολες ε, για να ε, μπορείτε εύκολα να μετακινήσετε στην πόλη της Βενετίας κύριε Πρόεδρε. Μία τελευταία παρατήρηση. Ένα σχόλιο που έκανε ο Γκέρτ για τα κρουαζιερόπλια που είναι ουσιαστικά πολυέροφα ε, λεωφορεία. Κοίταξε να δεις Τζόρτζ, εγώ έκλεισα διακοπές σε ένα κρουαζιερόπλιο. Αν πρόκειται για πολυέροφο λεωφορείο είναι πανάκριβο, πραγματικά. δεν ξέρω, ίσως πρέπει να περιγράψουμε στη Royal Caribbean και στην BNO και σε όλους αυτούς τους ανθρώπους ότι τα 850 εκατομμύρια δολάρια που έχουν επενδύσει δεν είναι τίποτα άλλο παρά μία επένδυση σε πολυέροφα Σχόλιο εκτός μικροφώνου του κ. Γραζεμπόφσκι. Δεν ξέρω, αλλά νομίζω ότι το τελευταίο κρουαζιερόπλοιο που πήγα δεν είχε πισίνα. Δεν ξέρω αν οι Γερμανοί με τα δικά τους τα λεωφορεία έχουν περισσότερο χώρο για πισίνα. Εγώ δεν είχα. Καλά περνάμε. Δεν βλέπω κάποια άλλη παρέμβαση. Η κυρία Βίτμαν τώρα για να θα σας απαντήσω αργότερα, κύριε Σίμψον. Euh, σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είπα και πριν από λίγο ότι στόχος μας είναι να έχουμε κοινέ αρχές σε όλα τα κράτη-μέλη, λαμβάνοντας βέβαια υπόψη τις ιτερότητες του κάθε κλάδου και λαμβάνοντας υπόψη και την προγενέστερη εμπειρία που έχουμε σε κάθε κλάδο. Όσον αφορά τις ιτερότητες του κάθε κλάδου θα πρέπει για το συγκεκριμένο να πω ότι μιλάμε για ένα κλάδο από το βασικό τμήμα, το βασικότερο ποσοστό του κύκλου εργασιών έχει να κάνει με τη μεταφορά εμπορευμάτων και πολλές φορές αναφερόμαστε εδώ πέρα σε λιμένες που δεν έχουν την κατάλληλη κατάρτιση, για τους, ε, την κατάλληλη υποδομή για την παροχή υπηρεσιών στους ε, επιβάτες. Επίσης, Έχουμε ορισμένα κράτη-μέλη τα οποία έχουν πολλούς και διαφορετικούς οργανισμούς για την επιβολή των ε, κανόνων και θεωρώ ότι τα κράτη αυτά έχουν και τα καλύτερα αποτελέσματα όσον αφορά την εφαρμογή των κανόνων. Θεωρώ λοιπόν ότι η πληθώρα οργανισμών δεν είναι απαραίτητα αρνητικό. Θα ήθελα για άλλη μια φορά να ευχαριστήσω τον ε, εισηγητή για την πολύ καλή αυτή έκθεση και την πολύ καλή συνεργασία που είχαμε. Θεωρώ ότι η έκθεση αυτή αποσαφηνίζει ορισμένα στοιχεία της πρότασης Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Γίνεται μια ευθυγράμμιση μάλιστα της διατύπωσης που χρησιμοποιείται. Θα ήθελα να διευκρινίσω κάποια πράγματα στα πλαίσια συζήτηση που έγινε. Η ε, υποχρέωση πληροφόρησης, ενημέρωσης, αρρωγής, αποζημίωσης είναι ανεξάρτητες από τους λόγους της καθυστέρησης ή τους λόγους προκαλούν ένα πρόβλημα. Μόνο στην περίπτωση της αποζημίωσης έχουμε συσχετισμό με τους συγκεκριμένου λόγους προκάλεσαν το πρόβλημα. Και κάτι ακόμα σε σχέση με το ερώτημα που ε, τέθη προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ναι, όντως τα ferry boat στους, ε, στα ποτάμια, στις πλωτές μεταφορές καλύπτονται εφόσον οι πλωτές εσωτερικές μεταφορές προβλέπονται στην πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστώ. Και όπως ξέρετε, οι εσωτερικές ε, ποτάμιες ε, μεταφορές περιλαμβάνουν και ε, τις λίμνες, οπότε μην ανησυχείτε, μπορείτε κάλλιστα να έρθετε στη Βενετία. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Θα σας βάλουμε στη γόνδολα και θα σας βυθίσουμε. Ο κύριος Τεσενέ. Σας ευχαριστώ, ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους για την ε, παρεμβάσεις τους. Περνώντας τώρα στη φάση των τροπολογιών θα πρέπει να καταφέρουμε να συγκλίνουμε κάπως τις απόψεις μας σε σχέση με τις προτάσεις που ακούστηκαν για τις κλιματικές, για τα κλιματικά προβλήματα που μπορούν να προκύψουν ή για τις εξαιρετικές συνθήκες που μπορούν να ισχύουν σε κάποιες χώρες. Αλλά με την καλή συνεργασία των σκεδών εισηγητών πιστεύω ότι θα καταφέρουμε να βρούμε την κατάλληλη ισορροπία, την πιο ικανοποιητική ισορροπία. Σας ευχαριστώ. Now we have a five minute break and then we have... Διάλειμμα 5 λεπτά και μετά ε, περιμένουμε την κυρία Τσικάου η οποία θα έρθει και θα ξεκινήσουμε με το επόμενο θέμα. Τελευταίο θέμα. You can light your cigarette and then and that will be more than enough. Ανάψτε το τσιγαράκι σας κύριε Γερζεμπός. Elle arrive, deux minutes.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 Okay. Ωραία λοιπόν, μπορούμε να συνεχίσουμε. πουντο 28-29 all'ordine del Σημείο 29 της μερίσιας διάταξης. Ok. Όροι που πρέπει να πληρούνται για την άσκηση του επαγγέλματος στο δικού μεταφορέα. Η συγκήτρια η κυρία Σίλβια Αντριάννα Τσικάου. Έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και να ευχαριστήσω πολύ και τους συναδέλφους που έχουν μείνει στην αίθουσα και ενδιαφέρονται για τη συζήτηση για το θέμα αυτό. Πιστεύω είναι πολύ σημαντικό να ξεκινήσουμε με το μήνυμα ότι έχουμε άλλες δύο ε, εκθέσεις οι οποίες αφορούν στο θέμα αυτό. Μία έκθεση του κυρίου Γκρός και τη δική μου. Και έχουμε και τα στοιχεία από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από το Συμβούλιο. και είναι πολύ ευνοϊκό το γεγονός ότι Το θέμα που προτάθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι κάτι το οποίο έχει ήδη ε, γίνει δεκτό από το Συμβούλιο και ε, θεωρώ ότι υπάρχουν κοινέ απόψει οι οποίες θα αντικατοπτρίζονται και στην τελική εκδοχή της έκδοση. Θα ήθελα να αναφέρω επίσης και το γεγονό ότι για κάποια από τα θέματα τα οποία έγιναν αποδεκτά και από το Συμβούλιο υπάρχουν ε, διστάμενες απόψεις και η έκθεσή μου ουσιαστικά είναι μια απάντηση ε, και προς υποστήριξη της θέσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και μια προσπάθεια να επισημάνουμε τις σημαντικές πτυχές. Υπάρχουν και κάποιες ε, τροπολογίες που αφορούν στο θέμα αυτό. Νομίζω ότι οι βασικές ε, διαφορές που έχουμε με το Συμβούλιο έχουν να κάνουν με το χρονοδιάγραμμα που προβλέπεται για τα ηλεκτρονικά μητρό, για την εφαρμογή ε, σε εθνικό επίπεδο και τη διασύνδεσή του σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το Συμβούλιο ήθελε ένα πάρα πολύ χαλαρό χρονοδιάγραμμα, ενώ το Κοινοβούλιο σε πρώτη ανάγνωση θεώρησε ότι τόσο οι πολύ σοβαρές παραβιάσεις όσο και οι σοβαρές παραβιάσεις θα πρέπει να ισχύσουν αυτή τη στιγμή σε εφαρμογή και ο κανονισμός. Μιλήσαμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και προσπαθήσαμε να ε, έχουμε ένα χρονοδιάγραμμα το οποίο θα έχει μια κάποια ευελιξία αλλά ε, δεν θα είναι τόσο ελαστικό όσο ήταν η πρόταση του Συμβουλίου. Και το Κοινοβούλιο εξακολουθεί να υποστηρίζει αυτή την άποψη. Υπάρχει και κάποιες μικροτεχνικές λεπτομέρειες. Ε, Παραδείγματο χάρη το Συμβούλιο ζήτησε να υπάρχουν και κάποιες διασφαλίσεις ε, για τις επαγγελματικές δεξιότητες. Ε, νομίζω ότι το Κοινοβούλιο μπορεί τελικά να τα δεχτεί αυτές τις διασφαλίσεις. Και υπάρχουν και κάποια στοιχεία τα οποία ε, θελήσαμε να τα συζητήσουμε με το Συμβούλιο, διότι φαίνεται ότι υπάρχουν μεγάλες διαφορές απόψεων ε, με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Για να μπορέσουμε όμως να δραστηριοποιηθούμε στην αγορά των μεταφορών, θα πρέπει να υπάρχει μία έγκριση για πρόσβαση στο επάγγελμα, αυτό αναφέρεται και στο έκθεσή μου, και επίσης θα πρέπει να υπάρχει και μία άδεια για την πρόσβαση στην αγορά. Αυτά είναι στοιχεία τα οποία αναφέρονται και στις ε, δύο εκθέσεις, ε, και στην έκθεση του κυρίου Γκρός και στη δική μου για τους επιβάτες. Το Συμβούλιο πρότεινε τα κράτη-μέλη να μπορούν ε, να περιορίσουν τη διάρκεια ισχύως της έγκρισης και για να μπορέσουμε να μειώσουμε τη γραφειοκρατία που αντιμετωπίζουν αυτές οι εταιρείε οδικών μεταφορών, ε, η έγκριση αυτή θα πρέπει να έχει μια διάρκεια 5 ετών, ώστε να μπορούν και οι αρμόδιες αρχές να διαπιστώσουν ε, αν πληρούν τα κριτήρια τα οποία ε, καθορίζει ο κανονισμός οι επιχειρήσεις αυτές και αν διαπιστώνουν ότι υπάρχει κάποιο συγκεκριμένος κίνδυνος θα μπορούσαν να κάνουν και κάποιους ε, σχετικούς ελέγχους. Το Συμβούλιο πρότεινε τα κράτη-μέλη να μπορούν να περιορίσουν τη διάρκεια ισχύω της εξουσιοδότησης της άδεια αυτής και θέλησε να εισαγάγει ένα κείμενο για το οποίο εγώ θα κάνω μία τροπολογία και θα ζητήσω τη διαγραφή του. Ε, αυτή τη στιγμή μια επιχείρηση θα μπορεί να ε, ζητήσει εξουσιοδότηση. Ε, θα πρέπει ο φορέας να μπορεί, ο μεταφορέας να μπορεί να λάβει και κοινοτική ε, έγκριση θα πρέπει να υπάρχει το θέμα της ε, πρόσβασης στο επάγγελμα, θα πρέπει να υπάρχει ε, πρώτερη έγκριση για την ε, αδειοδότηση στο επάγγελμα αυτό θα πρέπει να γίνεται, αλλά για την πρόσβαση στην αγορά θα πρέπει να ισχύουν τα όσα λέει και ο κύριος Γκρός. Και νομίζω ότι θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη αυτό το στοιχείο. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θέλει να επανεισαγάγει τη σημασία του να παρουσιάζονται, ε, να υπάρχουν ε, τα έγγραφα στην έδρα τους, ε, τα υπογεγραμμένα έγγραφα και εγκεκριμένα, Και επίσης το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ήθελε να περιλαμβάνονται και, τις, και οι μη εμπορικές υπηρεσίες οι οποίες αποκλείονται από τον κανονισμό αυτούς ε, τον κανονισμό αυτό, αλλά υπάρχει διαφορά απόψεων μεταξύ της θέσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Το Συμβούλιο θέλει να επανεισαγάγει αυτές τις εξαιρέσεις για τις εθνικές μεταφορές ε, ή για μεταφορές οι οποίες γίνονται σε, σύντομο, σε σύντομη απόσταση. Αρχικά το Κοινοβούλιο ήταν ε, κατά και θέλησε να συμπεριλάβει για κάποιες τροπολογίες για να επανέλθει η θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να συμπεριληφθούν αυτά στον κανονισμό. Θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ το Συμβούλιο που είναι παρόν εδώ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τους εκπροσώπους ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που είναι παρόντες εδώ. Κάναμε κάποιες ε, συναντήσεις με τους κοιόδης εισηγητές και θεωρώ ότι αυτά ήταν ιδιαίτερα θετικά διότι μπορέσαμε να αναπτύξουμε και κάποιες μελλοντικέ ε, προτάσεις για συμβιβαστικές τροπολογίες για το τελικό κείμενο. Περιμένω ε, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τη δική σας άποψη και πιστεύω είναι πολύ σημαντικό να σας πω ότι υπάρχει επιθυμία να επιταχύνουμε τη διαδικασία και να ε, να καταλήξουμε σε μια κοινή θέση. Αυτό νομίζω ότι ενδιαφέρει όλους μας, ε, διότι υπάρχει μεγάλο συμφέρον για αυτή τη συγκεκριμένη δραστηριότητα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριο Γερζεμπόφσκι. Ευχαριστώ να ευχαριστήσω και τη συνάδελφο εξ ονόματος της ομάδας μου για τις συζητήσεις με το Συμβούλιο και τη δέσμευση που επέδειξε. Ξέρω ότι δεν είναι απλά τα πράγματα. Ο συνάδελφος Γκρό ε, στη δική του έκθεση αναφέρθηκε ήδη για την έκθεση, στην έκθεση να Αναφέρω ένα στοιχείο θα ήθελα. Ο συνάδελφος Γκρός όπως και η δική μου ομάδα θεωρούν ότι είναι πάρα πολύ σημαντική η αυστηρή ρύθμιση σε ό,τι αφορά την ελευθερία εγκατάστασης. Αυτό το φαινόμενο των εταιριών γραμματοκιβώτιου θέλουμε να το πατάξουμε. Γι' αυτό πραγματικά όταν αναφέρεται μία έδρα θα πρέπει να υπάρχει έδρα, όχι να υπάρχει μόνο ένα γραμματοκιβώτιο. Το συζητήσαμε με αυτόν, ελπίζω να μπορείτε να τα βρείτε. Θέλουμε σε κάθε περίπτωση να αποτρέψουμε αυτές τις εικονικές επιχειρήσεις που δεν ε, βρίσκονται πραγματικά εκεί που λένε ότι βρίσκονται για φορολογικούς σκοπούς. Και είμαι βέβαιος ότι σωστά θα αντιμετωπίσετε μαζί με τον κύριο Γκρός. Κυρία Τικάου, σας ευχαριστώ. Η κυρία Λέχτεμπεργκερ. ευχαριστώ. Θα είμαι σύντομη. Συμφωνώ με αυτά που είπατε για τις εικονικές επιχειρήσεις. Δεύτερο στοιχείο. Στο ηλεκτρονικό αυτό μητρό θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να επιμείνουμε σε θέματα συμβατότητας. Γιατί αν δεν διασφαλιστεί το θέμα αυτό, θα καταλήξουμε σε ένα νεκροταφείο ουσιαστικά δεδομένων που δεν θα μας βοηθήσει σε τίποτα. Θα πρέπει κάπως να προσπαθήσουμε να το διασφαλίσουμε. Δεύτερο θέμα, σε ό,τι αφορά την ισχύ των αδειών και αυτή η προσέγγιση του Συμβουλίου. Κατά κάποιο τρόπο το καταλαβαίνω, ως ένα βαθμό, για το authorization. Γιατί τα κράτη-μέλη φυσικά θέλουν να είναι σε θέση να αντιδρούν στα προβλήματα. Αυτές οι αντιδράσεις όμως για να είμαστε ειλικρινεί, θα πρέπει να μπορούμε να τις διασφαλίσουμε και να τις ελέγχουμε. Δεν λύνεται αυτό με αδειοδότηση, αλλά με ελέγχου. Το πρόβλημα λοιπόν που αντιμετωπίζουμε είναι ότι τα κράτη-μέλη προβαίνουν σε ενστάσεις, αλλά όταν πρόκειται για την ίδρυση ελεγκτικών αρχών προκειμένου στοχοθετημένα να ανταποκρίνονται σε περιπτώσεις παραβιάσεων, όχι μετά από πέντε χρόνια σε ένα γενικό πλαίσιο, ε, τότε διστάζουν. Γι' αυτό λοιπόν θα προτιμούσα στοχοθετημένη αντίδραση σε προβλήματα μέσω ελέγχου σε περίπτωση ατασταλιών. Και σε αυτή την περίπτωση θα μπορεί να καταργηθεί, να αποσυρθεί μια άδεια και έτσι επιλύεται το πρόβλημα. Δεν θεωρώ ότι η χρησιτομή, δηλαδή είναι ο περιορισμός αλλά ο έλεγχος. Ίσως να χρειάζεται και κάποιος περιορισμός και βλέπω ότι διαφέρει η πραγματικότητα στα διάφορα και πρόκειται για ένα μήνυμα που αποστέλουμε ότι το θέμα αυτό εξακολουθεί να είναι αμφιλεγόμενο. Θα πρέπει να υπάρχει έλεγχος για να εξασφαλίσουμε ποιότητα αναφορικά με αυτά τα οποία αδιαφωτήθηκαν. Θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται. Δεν είναι δυνατόν, για παράδειγμα, να υπάρχει μια εταιρεία ταξί και να λέμε «Α, ο αδερφός μου ε, συμμετείχε στις εξετάσεις και πέρασε». Δεν είναι δυνατόν. Αυτές λοιπόν είναι οι δύο οδοί για να πετύχουμε το στόχο μας. Αναφερόμενοι στο στόχο μας αυτό σε ό,τι αφορά και την ε, πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα πρέπει να επιμείνουμε σε θέματα ελέγχου. Κύριε Σμίτ από την Επιτροπή. Ja, Dank, ähm, Herr Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Το σχέδιο κανονισμού για την άσκηση του επαγγέλματος αποτελεί ένα σημαντικό τμήμα του Road Package. Και χαίρεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που η συζήτηση μεταξύ Συμβουλίου και Κοινοβουλίου σημειώνει τόσο καλή πρόοδο. Γιατί προφανώ για μα είναι πάρα πολύ σημαντικό το στοιχείο των ελεκτικών μητρώων. Αυτό αποτελεί την κοινοτομία στο νέο αυτοκείμενο κανονισμού. Και με τον ελεκτικό αυτό μητρό θα είναι δυνατόν οι παραβιάσει οι οποίε γίνονται από επιχειρήσεις να καταστούν διαφανείς και μάλιστα διασυνεριακά γιατί σήμερα τι γίνεται στα εθνικά σύνορα πολλές φορές σταματάει. Η κατάσταση και οι αρμόδιες αρχές δεν γνωρίζουν καν τι κάνει μια επιχείρηση εκτός της επικράτειάς τους. Γι' αυτό λοιπόν είναι μεγάλη αυτή η πρόοδος το γεγονός ότι συμφωνεί το Συμβούλιο με το Κοινοβούλιο για τα ηλεκτρονικά μητρώα αυτά. Υπάρχουν κάποιες λεπτομέρειες όπως το άνοιγμα κάποιων τομέων ε, του Μητρώου αυτού για το ευρύ κοινό. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει να διτάξει κάτι, αλλά θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι δεν είναι αυτός ο βασικός σκοπός του Μητρώου. Ο βασικός σκοπός του Μητρώου είναι να ε, υπάρχει δυνατότητα συνεργασίας μεταξύ των εθνικών αρχών, αλλά υπάρχει και ένα επιπρόσθετο όφελος, γιατί όχι. Δεν είναι και το Συμβούλιο από ό,τι καταλάβαμε. Το Συμβούλιο όμως δυσκολεύεται σε ό,τι αφορά την εφαρμογή μας. Λέει σαφώς το Συμβούλιο ότι χρειάζεται πιο πολύ χρόνο από αυτό που προδιαγράφουμε εδώ στις Βρυξέλλες, το Κοινοβούλιο για παράδειγμα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό πρέπει πλέον να το αποδεχτούμε. Και θα πρέπει επίσης να σκεφτούμε ότι η επιμήκυνση των συζητήσεων θα αναβάλει ακόμα περισσότερο την εγκατάσταση των συστημάτων αυτών ηλεκτρονικού μητρώου. Αλλά θεωρώ ότι είναι καλό ως ιδέα. Τώρα, τα στοιχεία τα οποία ανέφερε η κυρία Τικάου. Καταρχάς, σε ό,τι αφορά, την διάρκεια ισχύω της άδειας, Να κάνουμε μία διάκριση. Ο κανονισμός αυτός αφορά τους όρους για την πρόσβαση σε ένα επάγγελμα. Δεν μιλάμε για άδεια, αλλά για το ποιοι είναι οι τέσσερις όροι οι οποίοι πάντα θα πρέπει να πληρούνται. Και θέλουμε αυτοί οι τέσσερις όροι και ο νέος όρος είναι ο όρος της εγκατάστασης, έχουν εισηχθεί σε αυτός ο όρος, αυτά θα πρέπει διαρκώς να ελέγχονται από τις αρμόδιες αρχές. Αν διαπιστωθούν ατασταλίες, θα πρέπει να δραστηριοποιηθεί λοιπόν η ηλεκτρική αρχή. Εμείς θεωρούμε και γι' αυτό έχουμε και το Μητρό ότι θα πρέπει να προκύπτει αυτό από το Μητρό. Μας λένε τα κράτη-μέλη ότι οι όρους υπάρχουν καταστάσεις όπου σωστό θα ήταν καταρχάς να περιοριστεί η διάρκεια ισχύω. Για παράδειγμα σε ό,τι αφορά νέες προσβάσεις, κάποιος που ξεκινάει με ένα επάγγελμα, ότι σκόπιμο θα ήταν να δίδεται άδεια για ένα-δύο έτη και μετά εφόσον αξιολογηθεί ότι καλά τα πήγε, να επιμεκυνθεί, να παραταθεί η άδεια αυτή. Εμείς μπορούμε να επιτρέψουμε αυτή την ευελιξία στα κράτη-μέλη. Δεν μιλάμε, δεν υπάρχει αναφορά σε μέγιστο, σε μέγιστη διάρκεια. Λέμε ότι τα κράτη-μέλη μπορούν, may, να ορίσουν τη διάρκεια. Και νομίζουμε ότι αυτό μπορούμε να το αποδεχτούμε. Επίσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί πάρα πολύ σημαντικό το φαινόμενο των ε, εικονικών επιχειρήσεων να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά και χαιρόμαστε που και το Κοινοβούλιο συμφωνεί προς αυτή την κατεύθυνση για την κατάρτιση κατάλληλων κριτηρίων. Νομίζω ότι αυτά είναι εν συντομία. Αυτές είναι οι θέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, για αυτό το πολύ σημαντικό πακέτο. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους ε, για τα όσα είπαν και τους κοιόδης συγητές με τους οποίους έχουμε ένα πάρα πολύ επικοδομητικό διάλογο. Για τις προτάσεις του κυρίου Γερζεμπόφσκι. Ναι, όντως επανήλθαμε με μια τροπολογία για να μπορέσουμε να υποστηρίξουμε τη θέση του Κοινοβουλίου σε πρώτη ανάγνωση, για να έχουμε την βασική έδρα των ε, εγγράφων και το γεγονός ότι η επιχείρηση θα πρέπει να μπορεί να πει πού βρίσκονται σταθμευμένα τα οχήματα που δεν βρίσκονται σε κυκλοφορία. Η τελική εκδοχή ήταν αυτή που εγκρόηθηκε και από το Κοινοβούλιο σε πρώτη ανέγνωση και ήταν πολύ πιο ευέλικτη από κάποιες τροπολογίες που κατατέθησαν που ήταν από πλευρά μου ως εισηγήτρια και έλεγα ότι το θέμα της στάθμευσης θα πρέπει να ρυθμίζεται από τους φορείς. θέλουμε να στηρίξουμε τη θέση της, ε, του Κοινοβουλίου σε πρώτη ανάγνωση για να μπορέσουμε να συμπεριλάβουμε αυτά τα στοιχεία και τα δικαιώματα των επιχειρήσεων σε αυτή την περίπτωση. Τώρα για τα σχόλια της κυρίας Λίχτεμπέργκερ. Πρέπει να σας πω ότι συζητήσαμε και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και με το Συμβούλιο και για να υπάρχει αυτή η σαφήνεια για τη συμβατότητα μεταξύ των ηλεκτρονικών μητρών η δομή των στοιχείων και τα στοιχεία που σχετίζονται με την αλλαγή των δεδομένων θα πρέπει να προκύψουν μέσω απόφασης. Θα πρέπει να υπάρχει ένα επίσημο έγγραφο και ένα, χωρίς να υπάρχει επίσημο έγγραφο τα κράτη-μέλη ε, θα μπορούν να πρέπει να τηρήσουν αυτά τα ελάχιστα όρια και από εκεί και πέρα να επεκταθούν σε εθνικό επίπεδο. Αλλά θα πρέπει να υπάρχει πρώτα ένα ελάχιστο όριο το οποίο θα διευκολύνει αυτή τη διαλειτουργικότητα. Όσον αφορά τώρα την ισχύ των εξουσιοδοτήσεων, εγώ είμαι της άποψης ότι θα πρέπει να είναι λίγο περιορισμένη. Θα πρέπει να έχουμε ένα μέγιστο των 5 ετών. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε πρώτη ανάγνωση είχε υποστηρίξει αυτή τη θέση, η οποία και εγκρίθηκε. Και όσον αφορά στις παρατηρήσεις ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, να ευχαριστήσω και τον κύριο Σμιτ για την καλή συνεργασία που είχαμε. Πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό τα κράτη-μέλη να κάνουν αυτή την επένδυση για να δημιουργήσουν αυτά τα ηλεκτρονικά μητρέα, διότι ε, θα είναι στοιχεία διάρκειας και είναι και ιδιαίτερα ευαίσθητα στοιχεία, τα οποία θα μπορέσουν να ωφελήσουν όχι μόνο τις αρμόδιες αρχές, αλλά και όλους όσους ενδιαφέρονται στον τομέα των οδικών ε, μεταφορών, ε, τους ε, οδικούς μεταφορείς, ε, αυτούς που μεταφέρουν εμπορεύματα. Υπάρχει το εμπιστευτικό κομμάτι στο οποίο θα μπορούν να έχουν πρόσβαση μόνο οι δημόσιες υπηρεσίες και αυτοί που έχουν έγκριση. Ε, το Κοινοβούλιο άλλωστε την υποστήριξε αυτή τη θέση στην πρώτη ανάγνωση. Επαναλαμβάνω, όσον αφορά την ισχύ των εξουσιοδοτήσεων, την ε, ισχύ λοιπόν των εξουσιοδοτήσεων πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό το θέμα αυτό. Όσον αφορά τώρα την πρόσβαση στο επάγγελμα, το να υπάρχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις οι οποίες θα πρέπει να επαληθεύονται πριν από την ε, γενική εξουσιοδότηση, αν θεωρείτε πέραν αυτών των πέντε ετών ότι υπάρχει κάποιος κίνδυνος από πλευράς επιχείρησης, μπορούν να υπάρχουν περαιτέρω έλεγχοι. Εδώ μιλάμε για την αγορά, ε, αναφέρεται και η έκθεση του κυρίου Γκρος στο θέμα αυτό. Όσον αφορά στα θέματα της αγοράς θα πρέπει να δούμε τα όσα ισχύουν στην έκθεση του κυρίου Γκρό. Όσον αφορά τώρα στην πρόσβαση στο επάγγελμα θα πρέπει να ε, βλέπουμε τι γίνεται με τον εφαρμοστικό κανονισμό για την ε, εξουσιοδότηση, για την πρόσβαση στο επάγγελμα του οδικού μεταφορέα. Θα πρέπει να εισαχθεί ένα ηλεκτρονικό το να υπάρχει ένας ε, εθνικός αριθμός ε, μητρώου θα μπορέσει να διευκολύνει τους ελέγχους, θα μπορέσουν να γίνουν τι γίνεται με τις ε, διασυνδέσεις και θα πρέπει να είναι διασυνδεδεμένα μεταξύ τους όλα τα δίκτυα. Περιμένω με ενδιαφέρον λοιπόν τις τροπολογίες σας και θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη συνεργασία που είχαμε, την ιδιαίτερα αγαστή και ελπίζω να καταλήξουμε τελικά σε μια κοινή θέση. Σας ευχαριστώ πολύ. Πολύ καλά. Να σας υπενθυμίσω την προθεσμία για τις τροπολογίες 12 η ώρα 25 Φεβρουαρίου. Με αυτό ολοκληρώσαμε την συνεδρίασή μας. Αν δεν υπάρχουν άλλα σημεία στην ημερήσια διάταξη που δεν υπάρχουν, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την ε, πολύ καλή συνεργασία ή στο επανειδή, στο επόμενο επεισόδιο.